προσαρμογή για τι άμεσε ενισχύσει, όσον αφορά το 2015. Το λόγο έχει ο κύριος Συγητή, ο κύριο Σικέρσκι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Σήμερα συζητούμε την έγκριση της τοποθέτησής μας σε σχέση με το ποσοστό αναπροσαρμογής για το ημερολογιακό έτος 2015, έτος δημοσιονομικής πειθαρχίας όπως αποκαλείται, όπως και προβλέπεται και στο οριζόντιο ψήφισμα του Δεκεμβρίου του 2013. Στα πλαίσια της τελευταίας μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής, βασικός στόχος της διαδικασίας είναι η δημιουργία ενός αποθεματικού για την αντιμετώπιση κρίσεων, για την στήριξη της γεωργίας όταν προκύψει μια σοβαρή κρίση που θα μπορούσε να πλήξει είτε την παραγωγή γεωργικών πρότατων είτε τη διανομή τους. Το συνολικό ποσό για την ε, περίοδο 2014-2020 ήταν 8 δις που σημαίνει γύρω στα 400 περίπου εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Με την ε, εφαρμογή της δημοσιονομικής πειθαρχίας ε, στις άμεσες ε, πληρωμές για το ημερολογιακό έτος 2015 προετοιμάζουμε ουσιαστικά τον προπολογισμό της Ένωσης για το έτος 2016. Στο σχέδιο προπολογισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει 441,6 εκατομμύρια ευρώ για το σκοπό αυτό, ως αποθεματικό δηλαδή. Μετά τις αρχικές εκτιμήσεις για τις άμεσες ενισχύσεις και τις σχετικές δαπάνες, τις σχετικές με την ε, αγορά γεωρικών προϊόντων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι αρκετή η αναπροσαρμογή των άμεσων ε, ενισχύσεων σε ποσοστό που δεν είναι καν το 1,4%. Και θα πρέπει να επιμείνουμε στο ότι μόνο για τους αγρότες που έχουν λάβει πάνω από 2.000 ευρώ άμεσων ενισχύσεων ετησίως, ε, σε αυτούς μόνο εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία. Επίσης, επειδή Βουλγαρία, Ρουμανία και Κροατία δεν έχουν φτάσει στο ανώτατο ποσό, δεν ισχύει αυτή η αναπροσαρμογή, αυτή η μείωση. Σύμφωνα με τον κανονισμό, το ποσοστό αναπροσαρμογής θα εγκριθεί στο πλαίσιο συναπόφασης Κοινοβουλίου και Συμβουλίου μέχρι το τέλος Ιουνίου, 30 Ιουνίου. Μετά αμέσως λοιπόν από την υποβολή του σχετικού αιτήματο ε, προς ε, την Επιτροπή Γεωργικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, Επιτροπή Γεωργίας, εμείς αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε την ταχεία διαδικασία, την απλουστευμένη διαδικασία, όπως ε, προβλέπει το άρθρο 50 του κανονισμού, ο πρόεδρος ε, της Επιτροπής, ο υποφαινόμενος συγκεκριμένα, συνέταξε έκθεση χωρίς τροπολογίες. Μετά την έκθεση της έκθεσης στην Επιτροπή Γεωργίας, χωρίς τροπολογίες, δεν υπευλήθη καμία τροπολογία ούτε και για την ε, τρέχουσα συνοδολομέλειας Ελπίζω λοιπόν αύριο στη διάρκεια της ε, ψηφοφορίας να εγκρίνουμε το σχέδιο της Κομισιόν χωρίς τροπολογίες. και θα πρέπει και το Συμβούλιο, ε, όπως έχει βεβαιώσει γραπτός, με δήλωση του Συμβουλίου θα δεχθεί αυτή την πρόταση της Κομισιόν χωρίς τροπολογής. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε συνένεση ήδη στην πρώτη ανάγνωση εντό της προθεσμίας ε, που προβλέπεται. Οι τελευταίες αναταράξεις ε, λόγω του ρωσικού εμπάρκου και λόγω της κατάργησης του συστήματος ποσοστώσεων στον τομέα των γαλακτοκομικών δείχνει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει αυτό το αποθεματικό. Ιδίω αν λάβουμε υπόψη του περιορισμού ε, των ε, μηχανισμών παρέμβαση, των διαφόρων προγραμμάτων παρέμβαση που θεσπίστηκαν με την τελευταία μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική Πολιτική. Επίση βλέπουμε ότι και εξωτερικοί παράγοντε έχουν όλο και μεγαλύτερη επιρροή. Η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου, για παράδειγμα, και το πώ επηρεάζει και την ευρωπαϊκή γεωργία. Επομένως, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πείσω κανέναν εδώ στην αίθουσα για το πόσο ευαίσθητος είναι ο τομέας της γεωργίας. Διότι εξαρτάται από το κλίμα, τις καιρικέ συνθήκες, την κερδοσκοπία, ε, τις διεθνείς αγορές και διεθνή συμβάντα. Επομένως, αν λάβουμε υπόψη ε, τις ε, παραθέσεις που προέκυψαν πέρυσι, βλέπουμε ότι πλέον επανέρχονται κονδύλια στον γεωργικό προπολογισμό και εκεί πρέπει να παραμείνουν για να αντιμετωπιστούν ε, οι επιπτώσεις της κρίσης. Πρέπει να υπογραμμίσω ότι το αποθεματικό αυτό αποτελείται από κονδύλια που προορίζονται αποκλειστικά για τη γεωργική πολιτική. Οι αγρότες για πάγωμα κάποιων πληρωμών, κάποιων ενισχύσεων ή εν μέρη δεν τους χορηγήθηκε αυτή η ενίσχυση, μπορούν πλέον να ξαναπάρουν αυτά τα κονδύλια. Επανέρχεται στο αποθεματικό. Ουσιαστικά το αποθεματικό είναι οι γεωργοί που το φτιάχνουν. Ευχαριστούμε και τώρα λόγο στον Επίτροπο, τον κύριο Χόγκαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια πολύ σύντομη εισαγωγή. Δεν θα με μακρηγορήσω όπως ξέρετε, στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ έπρεπε να ορίζουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο ένα σύστημα ευρωπαϊκό για τις άμεσες πληρωμές. Η πρόταση για τη μείωση ήταν για να χρηματοδοτήσουμε το αποθεματικό για την κρίση ε, το 2016. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στήριξαν την πρότασή μας και ελπίζουμε να υπάρξει έγκαιρη έγκριση της πρότασης πριν το τέλος Ιουνίου. Πολύ σωστά το επισημαίνει και ο συγκεκριτής. Ευχαριστώ. Ehm, Πράγματι ήταν συντομότατο. Θα δώσω τώρα το λόγο στου ε, συναδέλφου οι οποίοι έχουν εγγραφεί στον κατάλογο αρχή γενομένη από τον κύριο Μισελ που Υπάρχει το λόγο για δύο λεπτά. Δεν έχει ακόμη φτάσει ο κύριος Νταντέν οπότε θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Ντάντσιλα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επειδή το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών πρέπει να προστατεύεται, σε περίπτωση μείζωνος κρίσης, που μπορεί να προκύψει για διαφορετικούς λόγους ή καταστάσεις, και που μπορεί να επηρεάσει την ε, παραγωγή ή τη διανομή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φέτος έκανε μια πρόταση αναπροσαρμογής των άμεσων γεωργούς. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό αναπροσαρμογής των άμεσων πληρωμών είναι 1,39-30-41% και αυτές οι πληρωμές αφορούν τις, ε, τα ποσά άνω των 2.000 ε, ευρώ. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα αποθεματικό για τη χρηματοδότηση με 441 εκατομμύρια ευρώ και αν συγκρίνουμε τον αριθμό αυτό με τα 300 εκατομμύρια τη προηγούμενη χρονιά, καταλαβαίνουμε ότι σε περίπτωση κρίση της γεωργικής, του γεωργικού τομέα θα μπορέσει να αξιοποιηθεί καταλήλω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια νέα πρόταση αναπροσαρμογής, θα κάνει μάλλον μια νέα πρόταση να αναπροσαρμογής του ποσού αυτού ε, τον Δεκέμβριο του 2015, αναλόγως με τα στοιχεία του Νεμβρίου 2015. Το Κοινοβούλιο μελέτησε τα στοιχεία αυτά και για το τέλος Ιουνίου θεωρούμε ότι ο κανονισμός αυτός μπορεί να εγκριθεί. Ιδάλλως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίσει διαφορετικά για το ποσοστό αναπροσαρμογής. Ως εκπρόσωπος των Ευρωπαίων πολιτών θεωρώ ότι πρέπει να σεβαστούμε τις προθεσμίες που έχουν προβλεφθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο λόγος στον κύριο Κούσμιουκ για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, παίρνω το λόγο εξ ονόματο της ομάδας ECR για τον κανονισμό αυτό σε σχέση με το ποσό αναπροσαρμογή των άμεσων ενισχύσεων όσον αφορά το ημερολογιακό έτο 2015 που θα καταβληθεί όμως το 2016. Θα ήθελα να σα πω ότι στηρίζει η ομάδα μα τη λύση αυτή και θα υπερψηφίσουμε. Ο καθορισμός αυτού του ποσού αναπροσαρμογής ε, και η δημιουργία αυτού του ε, αποθεματικού για το ημερολογιακό έτος 2016 με ποσό 441,6 εκατομμύρια ευρώ σημαίνει ότι το εν λόγω αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχει κρίση στον γεωργικό τομέα. Είναι δε προφανές ότι αφορά τις άμεσες ενισχύσεις ποσών άνω των 2.000 ευρώ και ότι τρεις χώρες εξαιρούνται της μείωσης. Ωστόσο, παρά τον καθορισμό αυτού του ποσού και τη θέση του αποθεματικού, σημαίνει ότι οι εθνικοί προπολογισμοί των κρατών μελών θα μειωθούν. Και σίγουρα είναι ρευστή η καιρή και η κατάσταση που βιώνουμε ή δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό να έχουμε αυτό το αποθεματικό. Έχουμε το ρωσικό εμπάργκο, Επιδεινώνεται η γεωργική αγορά σε πολλούς τομείς και σε πολλές χώρες, όπως την Ανατουγάλυπτος για παράδειγμα. Επίσης, όλο και περισσότερες αγωγέ έχουμε στην Ένωση γεωργικών προϊόντων τρίτων χωρών και όλα αυτά αυξάνουν τους κινδύνους και την ε, ανασφάλεια. Αυτό το αποθεματικό λοιπόν θα στηρίξει τους αγρότες και τις αγορές που θα πληγούν πιο άμεσα από αυτά τα ενδεχόμενα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μίλλορ για δυόμιση λεπτά έχει τώρα το λόγο. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, η κοινή αγροτική πολιτική τα τελευταία χρόνια όλο και πιο πολύ κινείται και εξελίσσεται προς την κατεύθυνση των ανοιχτών αγορών. Η κατεύθυνση μαζί με την αποσύνδεση των άμεσων επιδοτήσεων και ένα βήμα για την επιχειρηματικότητα των ε, επιχειρήσεων έχει βάλει μεγάλες προκλήσεις ε, στις επιχειρήσεις. Αυτός ο προσανατολισμός σημαίνει και πιο, ψηλά, πιο ψηλούς κινδύνους για τις οικογένειες των αγροτών. Ιδιαίτερα οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι πολύ παραπάνω από, από ότι απλά τα σημεία παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Αυτές οι οικογενειακές επιχειρήσεις διασφαλίζουν ε, εκατομμύρια θέσει εργασία και διατηρούν την πολιτιστική κληρονομιά τη υπαίθρου τη Ευρώπη. Και ο κοινωνικό ιστό που υπάρχει στα χωριά μπορεί να διατηρηθεί μόνο μαζί με τι οικογενειακέ αυτέ επιχειρήσει. Όπω για παράδειγμα οι εθελούσιες δραστηριότητες πυροσβέσης ή και άλλες φύσεως δραστηριότητες. Τα προϊόντα και οι δομές αυτές βασίζονται στην οικογενειακή γεωργία. Αυτοί είναι κάποιοι μόνο από τους λόγους για τους οποίους μία απλή οικονομία της αγοράς χωρίς ε, μηχανισμούς εξασφάλισης δεν μπορεί να διατηρηθεί και να υπάρξει. Καλωσορίζουμε λοιπόν την ίδρυση ενός ε, ταμείου έκτακτης ανάγκης. Αυτό το αποθεματικό υπήρχε ως τώρα ήδη. Αφαιρέθηκαν διάφορα μέσα και από 5.000 ε, ευρώ και πάνω άμεσες επιδοτήσεις. Αυτό το όριο λοιπόν θα μειωθεί πλέον. Για μας και για τις οικογενειακές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σαφές πού πάνε τα χρήματα αυτά και πώς τα μέσα αυτά τα οποία πηγαίνουν στο αποθεματικό θα χρησιμοποιηθούν και η σημερινή κατάσταση με το εμπάρκο της Ρωσίας καταδεικνύει ότι και οι πολιτικές αποφάσεις μπορεί να ασκήσουν πίεση στην αγορά. Πέρα από το επιχειρηματικό σκέλος. Και εδώ θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όχι μόνο τα χρήματα των οικογενειών και επιχειρήσεων, αλλά και μέσα από τον προπολογισμό. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Νταντάν στο μεταξύ έχει καταφτάσει και θα του δώσω λοιπόν το λόγο. Σας παρακαλώ να με συγχωρήσετε, αλλά πολύ κολλήσαμε στο αεροδρόμιο του Στρασβούργου προηγουμένως. Δεν υπήρχαν ταξί. Ούτε κούρσες. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, με αυτή την έκθεση ένας από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς της κοινή αγροτικής πολιτικής και ε, έχει να κάνει με την ε, ε, χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε τα προβλήματα του ρωσικού εμπάργκο και των συνεπειών που μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμα για τον όλο μηχανισμό που έχουμε προβλέψει. Ήδη είχαμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε στην Επιτροπή Γεωργίας και το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν μια κρίση που έχει διπλωματικά αίτια και έχει πλήξει τους γεωργούς, αυτή είναι τα θύματα στην αγορά φέτος, δεν θα πρέπει να ε, αντιμετωπιστεί του χρόνου με την σωστή διαχείριση των ε, άμεσων ενισχύσεων. Δεν φταίτε εσείς Επίτροπε, ούτε εσείς ε, είστε στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης, όμως αφορά ένα μέρος του σώματος των Επιτρόπων και το σύνολο της λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Οι γεωργοί περιμένουν από εμά να δράσουμε, γι' αυτό σας ζητούμε Επίτροπε όλα αυτά να τα μεταφέρετε. Ευχαριστούμε. Τώρα η κυρία Σένρα Ροντρίκες. Για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνούμε ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει ένα αποθεματικό για την περίπτωση κρίση. Ε, ταυτόχρονα όμω, πρέπει να θεσπιστούν σαφή κριτήρια για να γνωρίζουμε όταν υπάρχει τέτοια κρίση. Η κοινή γεωργική πολιτική όσο έχει αυτή τη στιγμή δημιουργεί συνεχώ κρίσει στον τομέα τη παραγωγή Σήμερα, την ώρα που μιλάμε σε πολλέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τομέα του γάλακτο. Ε, αντιμετωπίζει βαθύτατη κρίση η παραγωγή. Ορίστε. Δεν υπάρχει στα γαλλικά μετάφραση από ό,τι φαίνεται. Λύθηκε το ζήτημα. It's okay, so please continue. Sorry. Ωραία. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Μπορείτε να, να ξαναρχίσω από την αρχή ή να συνεχίσω.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 Όπω έλεγα λοιπόν, συμφωνούμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα αποθεματικό για περιπτώσει κρίση, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να θεσπιστούν σαφή κριτήρια για να γνωρίζουμε πότε προκύπτει κρίση. Η κοινή γεωργική πολιτική, όσο έχει αυτή τη στιγμή, προκαλεί βαθύτατε ε, κρίσει ε, μόνιμα ε, στον τομέα τη παραγωγή. Σήμερα, αυτήν την ώρα που μιλάμε, σε πολλέ χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων η χώρα μου, η Γαλλικία, οι παραγωγοί γάλακτος έχουν πιάσει πάτο. Οι τιμές κάτω από το κόστος παραγωγής. Οι επιχειρήσεις πάρα πολλές, ε, πολλούς ανεξόφλητους λογαριασμούς δεν έχουν πληρωθεί για το γάλα. Ε, πώς ε, ε, θα λύσουμε τα προβλήματα. Ναι, είναι η οικονομική στήριξη απαραίτητη. Αλλά θα πρέπει να έχουμε και μια δημόσια πολιτική για τον τομέα του γάρτος για να αποφύγουμε τέτοιε καταστάσει. Επίση, πιστεύουμε ότι οι κρίσει που προκαλούνται λόγω σφαλμένων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως αυτές που οδήγησαν ε, στο ρωσικό εμπάρκο θα πρέπει να αντισταθμίζονται με άλλα κονδύλια και όχι με τη στήριξη αυτού του αποθεματικού που είναι για τους γεωργούς, για τους αγρότες. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φερόν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε και κύριοι. Πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω ε, μια ομάδα αμπελουργών που έχουν έρθει από τη Βουργουνδία μαζί μας, μια μεγάλη, ε, μια ένδοξη ε, περιοχή για την παραγωγή ίνου ε, κύριε Επίτροπε, οι στιγμέ είναι δύσκολε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή στα γεωργικά ζητήματα ακολουθεί αυτοκτονική πολιτική. Ο κύριο Σούλτ και οι φίλοι του τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν προβλέψει κυρώσει κατά τη Ρωσία. Όμω, σήμερα ολόκληρη η Ήπειρο πλήττεται από τι πολιτικέ αυτέ προτεραιότητε. Και οι Γεωργοί είναι θύματα δύο φορές. Πρώτα απ' όλα από το ρωσικό εμπάργκο που έχει κοστίσει μόνο για τη Γαλλία. Μόνο για τη Γαλλία ακούσαμε ένα δις ευρώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σκαλίσει ε, και έχει βρει ε, ποσά από την γεωργική πολιτική για να αποζημιώσει δίθεν αυτούς τους γεωργούς. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αρθούν οι κυρώσεις και να μπορέσουν να επιβιώσουν οι γεωργοί να αναπνεύσουν και στην Ευρώπη και στη Γαλλία. Ευχαριστούμε. Η κυρία Εράς Καρσία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Σιγέρσκι για το έργο του ως εισηγητού για την έκθεση αυτή και κατά δεύτερον θα ήθελα να συγχαρώ και τον Επίτροπο εξ ονόματος ε, του Συνόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτή την πρόταση που διατηρεί το παθεματικό. Αυτό το οποίο θεσπίστηκε με την τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΑΠ Στόχο του εργαλείου αυτού είναι ε, να είναι διαθέσιμα κονδύλια για την αντιμετώπιση κρίσεων, ε, όταν βέβαια αυτέ είναι σοβαρέ, ε, αλλά 442 περίπου εκατομμύρια ευρώ δεν αρκεί ως ποσό. Αυτό συνεπάγεται περισσότερε προσπάθειε από του αγρότε που βλέπουν να μειώνονται οι άμεσε ενισχύσει για να καλυφθούν προβλήματα στην αγορά που θα μπορούσαν να είχαν καλυφθεί εάν χρησιμοποιούν τα περιθώρια του προπολογισμού. Και πολλές φορές ξέρουμε ότι δεν χρησιμοποιούνται αυστηρά και κυρικές δαπάνες σε αυτά τα κονδύλια. Έχουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία, ένα μηχανισμό που ε, μπορούμε να ε, χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε ε, για να λύσουμε προβλήματα τα οποία δεν οφείλονται όμως άμεσα στο γεωκοτομέα, όπως για παράδειγμα με το ρωσικό εμπάργο και έγιναν, έγιναν προσπάθειες να βάλει χέρι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το αποθεματικό ε, που είναι μόνο για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και ευτυχώς η πλειοψηφία του Κοινοβούλου ήταν κατά. Ε, πιστεύω ότι και τέτοιες κρίσεις και κατά το παρελθόν αλλά και σήμερα θα μπορούσαν να χρηματοδοθούν από άλλα κονδύλια σήμερα να ρωτήσω τι εγγύσει έχουμε ότι αυτό το αποθεματικό δεν θα χρησιμοποιηθεί εάν το ρωσικό εμπάρκο επιμηκυνθεί ακόμη περισσότερο και μετά το καλοκαίρι. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό το αποθεματικό θα πρέπει να είναι μήνυ ανέγκυχτο προς το παρόν για να μπορέσουμε να δώσουμε άχρηστη μια γρήγορα αποτελεσματική απάντηση ως Ευρώπη απέναντι σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει λόγω εγγενών εξελίξεων ε, στις γεωρικές αγορές, αλλά μιλάω μόνο για τις γεωρικές αγορές. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιούμε πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους. Και καταλήγω με αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Μπράραν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η ετήσια άσκηση αποθεματικού για κρίση στον γεωργικό τομέα βοηθάει στην προστασία των εσόδων των γεωργών σε περίπτωση ε, διακυμάνσεων των τιμών ή κρίσεων. Και αυτό είναι ένα δίκτυο προστασίας που προστατεύει από αναπάντηχα γεγονότα το αποθεματικό κρίση χρηματοδοτείται από τον φάκελο για τι άμεσε επιδοτήσεις. Αυτό είναι δίκαιο και λαμβάνει υπόψη ότι ο προπολογισμό που ήδη είναι βεβαρημένο δεν θα πρέπει να, δεν θα βρεθεί σε θέση να αναγκαστεί σε περίπτωση κρίση, να επιβαρυνθεί σε περίπτωση κρίση. Θα πρέπει να κοιτάξουμε πιο πολύ το δυναμικό διαχείριση κινδύνου τη ΚΑΠ και να δώσουμε πιο πολύ προσοχή σε ενδεχόμενα μερικά προβλήματα. Αντί να επικεντρωθούμε στην υποστήριξη εισοδήματο, θα πρέπει να εστιαστούμε στα ποσά τα οποία μένουν σε αποθεματικό για σε περίπτωση κρίσης φυσικών καταστροφών εμπάρκο. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη τις ε, ανάγκες του κλάδου για να μπορέσουμε με σωστό και σόφρονο τρόπο να δαπανίσουμε τις, ε, τα κονδύλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Βουτσικόφσκι για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε η μεγάλη αξία της Ευρώπης είναι η αλληλεγγύη, η αρχή της αλληλεγγύης. Ένας ε, για όλους και όλοι για τον έναν. Στο όνομα λοιπόν της αλληλεγγύης επιβλήθηκαν και κάποιες κυρώσεις στην Ρωσία γιατί αυτό προαπαιτούσε οι αξίες της Ευρώπης την αντίσταση στην ε, επέκταση της Ρωσίας, αλλά το σκέλος της αλληλεγγύης δεν λειτουργήσε επαρκώς. Γιατί οι Γεωργοί είναι αυτοί που πληρώνουν τα σπασμένα στις βαλτικές χώρες, στη Φιλανδία, στην Πολωνία. Οι Γεωργοί δεν έχουν να πουλήσουν τα μήλα τους, το γάλα τους στην Πολωνία. Ήταν πραγματικά τραματική η κατάσταση σε ό,τι τον κλάδο των ε, μήλων. Χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία σημείωσαν μεγάλες ε, απώλειες στα έσοδα ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ. Και οι αποζημιώσεις είναι σε επίπεδο εκατοντάδων ευρώ. Δεν είναι λοιπόν δίκαιη η κατανομή των ε, μέσων αυτών. Αυτές οι ετησίως καθοριζόμενες λύσεις ε, για αποθεματικό δεν χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό και διερωτώνται οι Γεωργοί. Πού χρησιμοποιούνται τα μέσα αυτά? Θα ήθελα λοιπόν να χρησιμοποιηθούν με σωστό τρόπο αυτά τα μέτρα. Ο κ. Γιάκοφτσης για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. κύριε Σιγητά. Να πω ευθύ εξ αρχής ότι στηρίζω τη δημιουργία αυτού του αποθεματικού κρίσης, διότι είμαι το πεπισμένος ότι ένα τέτοιο αποθεματικό είναι απαραίτητο για τους αγρότες σήμερα. Και αυτό δεν σχετίζεται μόνο με τη σημερινή κατάσταση με τη Ρωσία, που φυσικά και θα πρέπει να μας ενθαρρύνει στο να διαθέσουμε αυτά τα χρήματα, να έχουμε αυτό το αποθεματικό. Όμως, και η γενικότερη κατάσταση και η ανάγκη να προστατεύσουμε τους ε, αγρότες ε, είναι επιχειρήματα που συγχωρούν υπέρ της ε, δημιουργίας αυτού του αποθεματικού. Οι αγρότες μας είναι αντιμέτωποι με τεράστιες προκλήσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, κύριε Σιγητά, είναι καλή πρόταση για τη δημιουργία ενός τέτοιου αποθεματικού θα δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια στους αγρότες μας και θα μας δώσει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να επιδείξουμε αλληλεγγύη, κάτι αναγκαίο είναι άλλωστε και ένας από τους ακρογωνίους λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αλληλεγγύη. Λέμε για ότι η Κροατία, η χώρα από την οποία κατάγομαι, δεν θα ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό. Αλλά θα συμμετέχει ε, το 2022 πλήρως. Εγώ θα ήθελα να μην προκύψει κάποιο πρόβλημα για τους δικούς μας γεωργούς. Ούτε όμως και για τους ε, γεωργούς από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία που αυτοί θα συμμετέχουν από του χρόνου. Η Κροατία όμως, όπως είπα, από το 2022. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι και οι αγρότες των χωρών αυτών θα είναι επιλέξιμοι για κονδύλια από αυτό το αποθεματικό, γιατί και αυτοί πλήττονται από τις ρωσικές κυρώσεις και το ρωσικό εμπάργο. Έχουμε και εμείς στην Κροατία πρόβλημα με την ε, εξαγωγή μανταρινιών για παράδειγμα. Πώς θα συμπεριλάβουμε λοιπόν τους ε, αγρότες ε, όλων των χωρών σε αυτό το επιθεματικό. Ευχαριστούμε κύριο Φλάνναγκαν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ με την ιδέα να υπάρχει αποθεματικό για να βοηθήσουμε τους Γιώργους, ούτως ή άλλως. Είναι λίγο λυπηρό που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει χωροφύλακας του διεθνού προσκυνίου και αυτό πλήττει του Ευρωπαίου γεωργού. Από ό,τι καταλαβαίνω, αποτελέσματα δεν έχουμε. Και καλό θα ήταν να γίνει κάτι, ε, αλλά όχι ότι να είναι μόνο και μόνο για να φανεί ότι δρούμε. 35 ε, εκατομμύρια έχουν χάσει οι Ιρλανδοί γεωργοί και εκατοντάδε εκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη. Τι πετύχαμε. Ε, ξεκονόμηση για πραγματικέ κρίσει δεν έχουμε κάνει. Στην Ιρλανδία, ε, βάσει τη ΚΑΠ, έχουμε ήδη ένα αποθεματικό. 80% τη χρηματοδότηση τη ΚΑΠ ε, πηγαίνει στου πλουσιότερου γεωργού. Γιατί υποτίθεται ότι αυτοί πρέπει να προστατεύονται. Οι μικροί γεωργοί και οι οικογενειακέ εκμεταλλεύσει, καληνύχτα σα στη χώρα μου. Αυτού όμω πρέπει να βοηθούμε επί τη ουσία. Ευχαριστούμε ο κύριο Μπούντα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Σιγητά, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι, είναι απαραίτητο αυτό ο μηχανισμό για να έχουμε βιώσιμη και αποτελεσματική γεωργία. Γι' αυτό χαιρετίζω την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίω ε, όσα είπε ο Επίτροπο Χόγκαν για να προβλέψουμε καλύτερες συνθήκες για τον γεωργικό τομέα. Θα πρέπει να δώσουμε στους γεωργούς τη δυνατότητα και να πληρώνεται το ποσοστό αναχρωματοδότησης για τις άμεσες πληρωμές, ε, για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήματα το 2015 χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τι ε, πληρωμές έχουν γίνει ε, προηγουμένως τα κράτη-μέλη μπορούν να ε, καταβάλουν τις πληρωμές αυτές με καθυστέρηση, πρόθεσμα δηλαδή, εφόσον τα αιτήματα έχουν υποβληθεί εγκαίρως. Πάντω, καλώ κάνουν διάκριση μεταξύ των κρατών, δεν κάνουν διάκριση μεταξύ των κρατών μελών για τις άμεσες πληρωμές και οι ευρωπαϊκοί γιατί αυτό θα δημιουργούσε μεγάλη ένυψη ισορροπία. Δεν μπορεί να λαμβάνουν ακριβώ το ίδιο ποσό οι Ρωμανοί Γεωργοί όμω, όπω και σε άλλε χώρε. Αυτό δεν είναι σωστό. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε έναν αποτελεσματικότερο μηχανισμό στο μέλλον για να αμφιδίσουμε τους γεωργούς και κάθε περιοχή να ε, λαμβάνεται υπόψη ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής του στον Ευρωπαίο, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Χώρο. Επίσης, θα πρέπει να βρεθεί μια γενικότερη ισορροπία μεταξύ των επιδόσεων των γεωργών, της προσβασιμότητας και της καμηλής τιμή των γεωργικών προϊόντων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη και να μην ξεχνάμε ότι όσα συμβαίνουν στη Ρωσία ε, πλήττουν την αγορά. Δεν είναι αρκετά δυνατή, οπότε χρειάζεται μια κοινή προσπάθεια για να βρούμε βιώσιμες λύσεις. Ε, ε, Ευχαριστούμε κύριο Ντενανό για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι αυθαίρετο αυτό ποσοστό του 1,39 για το 2016 φαίνεται εύλογο βάσει των στοιχείων που διαθέτουμε. Έτσι φαίνεται. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι να ορίσουμε σωστά τα ποσοστά. Το πρόβλημα είναι το δημοσιονομικό περιθώριο που έχουμε στι περιπτώσει των πιστώσεων. Αυτό ήθελα να το υπογραμμίσω. Ε, και μάλιστα στη γνωμοδότηση που έχω ετοιμάσει για την Επιτροπή Γεωργικών ε, Θεμάτων ε, για το 2016. Εκεί σε περιπτώσει μείζωνο κρίση πρέπει να χρησιμοποιούνται τα περιθώρια του κεφαλαίου 2 που υπάρχουν διαθέσιμα σε περίπτωση κρίσεων και ω αποθεματικά. Όπω υπόθηκε επανειλημμένω, οι κρίσει στο γεωργικό τομέα μπορεί να γίνουν σύνηθε φαινόμενο εξαιτία του εμπάργκο κατά της Ρωσίας. Αυτές οι απειλές είναι γνωστές σε όλους. Θα πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους γεωργούς που έχουν πληγεί και από το ρωσικό εμπάργκο και επειδή για τα οποροκυπευτικά σε όλες τις περιφερειές υπάρχει πρόβλημα και να μην ξεχνάμε και το θέμα της αγοράς του γάλακτος με τις νέες ποσοστώσεις και αυτό μπορεί να απειλεί σε πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις και εκτινοτροφικές μονάδες και στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ευχαριστώ. Ashworth, ένα λεπτό. Uh, Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνω και εκτιμώ την πρόθεση της αλληλεγγύης και του επιθυματικού για την αντιμετώπιση της κρίσης. Παρά το γεγονός ότι δεν το υποστηρίξει η ομάδα μας στην αρχή, έχουμε την αίσθηση ότι μπορεί να υπάρχει καλύτερος και πιο δίκαιος τρόπος να χρηματοδοτηθεί αυτή η διάταξη. Δεν έχω πρόβλημα να μειωθούν τα κατόφυλλα για τις ε, εισφορές, αλλά θα πρέπει να εκφράσω την ανησυχία μου για τον αντίκτυπο που θα έχει στους παραγωγούς στη δική μου χώρα. Πρόκειται για μια χώρα που λόγω των δομών της ε, έχει λιγότερες μεγάλες επιχειρήσεις από ότι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό τι σημαίνει ότι οι μεμονωμένοι παραγωγοί έχουν ήδη μεγάλο βάρος ε, και θα έχουν πολύ μεγαλύτερο μερίδιο του βάρους από ότι ο μέσος αγρότης. Αυτό για μια εισφορά σε ένα ταμείο το οποίο από πλευρά παράδοση πάντα αρνούταν και δεν ήθελε η κυβέρνησή του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο πρόεδρο. Και τώρα. Ο κ. Σαλή, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η εφαρμογή των διατάξεων που ορίζει ο κανονισμός για την παρακολούθηση της ΚΑΠ και η δημιουργία κανόνος για τις άμεσες επιδοτήσεις είναι σημαντικά στοιχεία στην διαδικασία κατάρτισης του προπολογισμού για το 2016 σύμφωνα με τον κανονισμό για την προστασία του γεωργικού κλάδου σε περίπτωση κρίσης το αποθεματικό για την κρίση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριληφθεί στο σχέδιο προπολογισμού είναι 441,6 εκατομμύρια ευρώ και η ρήτρα αναπροσαρμογή 1,39% που ελπίζουμε να υπολογιστεί σωστά και αυτό βασίζεται σε υπολογισμούς για άμεσες ενισχύσεις ε, σε ό,τι αφορά τα 2.000 ευρώ και δεν είναι συμπεριλαμβάνονται και κάποια κρατημέλη. Αυτό σημαίνει πιο, πιο λίγα χρήματα για τους γεωργούς και θα ήταν ένα καλό βήμα να γίνει αυτό σε μπορούσα φάση για την απλοποίηση των ε, αιτήσεων για τους μικρούς εκμεταλλευτές, για τους μικρούς γεργούς. Σε ό,τι αφορά τη σωστή εφαρμογή, υποστηρίζουμε την έκθεση σε ό,τι αφορά το 2015. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τάρασο, για ένα λεπτό έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Οι μικροί γεωργοί κτηνοτρόφοι από την Νότια Ευρώπη ζουν μόνιμα σε κατάσταση κρίσης εδώ και χρόνια. Ξέρετε από την Αστούρια ε, πόσο πωλείται το ένα λίτρο ε, γάλακτος 33 σέντ. Καλό είναι να έχουμε αυτό το αποθεματικό, όχι όμως και να ε, χαιρόμαστε τόσο πολύ. Δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα και μου είπε και ένας ε, πρόσφατα, ένας Γιώργος, δεν θέλω ελεημοσύνη, απλά θέλω να πάρω κάτι πίσω από το προϊόν το οποίο πολλώ για να ζω με αξιοπρέπεια. Το αποθεματικό σίγουρα ε, θέλει να δημιουργήσει συνθήκες για την αντιμετώπιση κρίσεων, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο παραγωγικό που θα προστατεύει ε, τα δημόσια αγαθά και όχι τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων. Το χρωστούμε στον κόσμο, ο οποίος πλήττεται τώρα από τις εσφαλμένες αποφάσεις. Το οφείλουμε στους πολίτες ε, να κοιτάμε ψηλά, να βάλουμε ψηλά τον πύχη. Ευχαριστώ. Κυρία Σχράιερ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, καταρχά θα ήθελα να πω ότι η πρόταση του εισηγητή με βρίσκει απόλυτα σύμφωνα γιατί το μποϊκοτάρισμα της Ρωσία έχει πλήξει σοβαρά τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Η εξαγωγή Ολλανδικών προϊόντων στη Ρωσία έχει μειωθεί κατά 30% και πλέον φέτος. Η οικονομική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σημαντική λοιπόν για το έτος αυτό για πολλές οικογένειες αλλά και για πολλούς ε, συνδεδεμένους τομείς και θα πρέπει λοιπόν να τηρηθεί σε ίδια επίπεδα. Τα πιο πολλά χρήματα πήγαν στα προκυβευτικά και στα γαλακτοκομικά, αλλά υπάρχουν και άλλοι κλάδοι και κοιτώ προς τον ε, Επίτροπο μίλησε για τον τομέα της παραγωγής χείρων που επλήχθησε σοβαρά στην Ολλανδία. Θα πρέπει λοιπόν η κρίση να έχει και θετικά αποτελέσματα. Να δούμε πώς μπορούμε να την ε, χρησιμοποιήσουμε με θετικό τρόπο. Και στο μέλλον θα πρέπει όλα τα μέσα από το Ταμείο για την Κρίση να μπορούν να χρησιμοποιούνται. Ξέρουμε ότι τα μέσα τα οποία δεν αξιοποιούνται επανέρχονται στην ε, καλλιέργεια, στους καλλιεργητές και στους παραγωγούς γάλακτος. Αυτό είναι καλό. Αλλά ζητούμε παράταση από τον Ιούλιο μέχρι 7 Αυγούστου για να δούμε και τους εθνικούς φακέλους, να δούμε και τους ε, τομείς που δεν έχουν ακόμα, δεν είναι ακόμα στην κρίση, γιατί κοιτώντα ας πούμε τους παραγωγούς της ντομάτας θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά. Ένα σημείο είναι σημαντικό. Είμαστε υπέρ της Ευρώπης των λιγότερων μικρών κανόνων και βλέπω ότι οι γεωργοί μας και οι καλλιεργητές μας δεν ξέρουν πώς να χρησιμοποιήσουν σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς τις δυνατότητες που έχουν. Και αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να το λύσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η... Ο κύριε Τρεπίκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Προφανώς έχουμε ανάγκη από ένα τέτοιο είδους εργαλείο για την αντιμετώπιση των, ε, της και για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κονδύλια προς όφελο των γεωργών. Ταυτόχρονα πρέπει να λάβουμε υπόψη το εξή. Είναι σημαντικό το αποθεματικό αυτό να χρησιμοποιηθεί ε, για το σωστό σκοπό προκειμένου να βοηθήσουμε τους γεωργούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το ξέσπασμα μιας κρίσης όπως αυτό που συνέβη με το ρωσικό εμπάργκο. Είναι σημαντικό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει σωστά το ρόλο της και γι' αυτό εμπιστεύομαι, πρέπει να πω, τον Επίτροπο Χόγκαν, ο οποίος θα ορίσει σαφείς όρους για τους δικαιούχους αυτού του Ταμείου. Δεν ε, μπορείτε δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι θα πρέπει να απευθυνθεί στους αυτούς δικαιούχους το αποθυματικό αυτό. Και επίσης να μην προκύψει ανταγωνισμό μεταξύ των γεωργών λόγω των διαφορών στα ποσά που θα πληρωθούν. Πιστεύω ότι πρέπει να εξαλείψουμε τις άμεσες πληρωμές γενικότερα. Ε, ε, ε, Øh, øh, Ο κύριο Ντόρμαν, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, σε όλε τι χώρε θεωρούμε το θέμα αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να συνεργαστούμε λοιπόν υπέρ των γεωργών. Δυστυχώ, όλοι το γνωρίζουμε ότι το 2016 θα είναι ένα έτος το οποίο ενδεχομένω να δημορφωθεί με πολύ δύσκολο τρόπο για τον κλάδο τη γεωργία Σε ό,τι αφορά και το εμπάρκο τη Ρωσία. Ε, γιατί αυτό ενδεχομένω να οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας. Και πώς μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε τον γεωργικό κλάδο, αυτό σίγουρα θα πρέπει να μα απασχολήσει και θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν να υπάρχουν κάποια μέτρα βοήθειας ε, ε, για του γεωργούς που πληρώνουν ε, μεγάλο τμήμα σε αυτές τις εποχές κρίση. αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με το ρωσικό εμπάργκο στο μέλλον. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το τύπημα της πολιτικής, του πολιτικού χαυγά μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας είναι πολύ υψηλό και το πληρώνουν οι γεωργοί. Και θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε νέες αγορές εξαγωγής για τα προϊόντα τα οποία παλιά πολλούνταν στη Ρωσία, γιατί η Ρωσία ήταν σημαντική αγορά για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και το ξέρετε όλοι άλλωστε ότι οι Δανείοι πολλούν μεγάλες ποσότητε χειρίου κρέατος. Εδώ λοιπόν έχουμε πληχθεί ιδιαίτερα και θα πρέπει να εξευρεθούν εναλλακτικέ αγορές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Δεν υπάρχει θέμα για την ανάγκη ύπραξη αποθεματικού για περίπτωση κρίση. Όμως η ΚΑΠ αυτή η ίδια είναι αίτιο κρίση Η τελευταία μεταρρύθμιση προκάλεσε σκανδαλώδεις ανισότητε μεταξύ των κατανομή των κονδυλίων και μεταξύ των χωρών, των παραγωγών και των γεωργών. Ο προσανατολισμό της αγοράς έχει οδηγήσει ε, εκατομμύρια μικρούς γεωργούς σε ε, αδιέξοδο. Εδώ βλέπουμε να μην υπάρχει σωστή παραγωγή, να καταστρέφονται γεωργικές μονάδες, να συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένα χέρια οι μεγαλύτεροι τομείς παραγωγής και μετά υπάρχει και η ανταγωνιστικότητα που όμως ε, για κάποιους σημαίνει ότι θα πάρουν τα διπλάσια, τριπλάσια ποσά ένα εκτάριο από ότι άλλοι. Έτσι είναι πολύ εύκολο να κάνει ανταγωνιστικό. Στην Πορτογαλία ε, χιλιάδε, δεκάδε χιλιάδε μικροπαραγωγοί ε, δίνουν μάχη για να επιβιώσουν, ε, για να μπορέσουν να έχουν μια ελάχιστη παραγωγή χωρί να καλύπτουν το κόστο όμω. Και αυτό ε, με 500 ευρώ που θα λάβουν για το, από την άμεση πληρωμή προφανώς δεν θα μπορέσουν να ξεπεράσουν την κρίση. Ευχαριστούμε ε, η κυρία Ριμπέιρο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ε, Επίτροπε, την τελευταία κρίση οι Ευρωπαίοι Γεωργοί έχουν μπει σε μια οικονομική πειθαρχία ε, που δεν τους επιτρέπει με το αποθεματικό που προβλέπει ο προπολογισμό να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που υποτίθεται θέλει να, ε, σώσει, να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει τα ποσοστά ε, κάτω των 2.000 ευρώ να έχουν και αυτά ένα ποσοστό αναπροσαρμογή κατάλληλο. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το κεφάλαιο που αφορά την γεωργία με συνεπείς προσπάθειες από όλες τις πλευρές και και να κοιτάξουμε συνολικά ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν είναι σωστά καταρτισμένο για να υπάρξουν νέε επενδύσει στον τομέα όπω απαιτείται. Αυτό το μήνυμα πρέπει να ακούγεται και από του παραγωγού μα, διότι οποιαδήποτε δημοσιονομική ενίσχυση προ τον τομέα θα πρέπει να μην οδηγήσει σε περικοπή των άμεσων πληρωμών προ του γεωργού που πάνω απ' όλα τα χρειάζονται. Ε, κύριε Επίτροπε, ε, υπάρχουν έκτακτε καταστάσει που απαιτούν όμω και έκτακτε αποφάσει. Ε, πρέπει λοιπόν οι Ευρωπαίοι, οι Ευρωπαίοι γεωργοί που απειλούνται και η επισητιστική ασφάλεια που απειλείται ταυτόχρονα να αντιμετωπιστούν υπό το φω του ρωσικού εμπάργκο. Είναι μεγάλη η κρίση στον τομέα και ακόμα ε, βλέπουμε του τριγμού από τι συνέπειε θα πρέπει τη μείωση των εισοδημάτων που είναι δραματική σε ορισμένε περιοχέ, όπω τι εξόχου απόκεντρε, να την αντιμετωπίσουμε. Απαιτούνται διπλωματικέ και πολιτικέ αποφάσει, γιατί τελικά τι οικονομικέ κυρώσει τι έχουν πληρώσει οι γεωργοί μα. Πώ αυτή η κρίση να ξεπεραστεί από τον τομέα, όταν βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αντιμετωπίζει άμεσα τι επιπτώσει τη κρίση. Τα κονδύλια δεν έρχονται από άλλον ε, τομέα, από άλλο κεφάλαιο του προπολογισμού. Και για τον τομέα του γάλακτος είδαμε ότι η παρέμβαση στην αγορά δεν έχει φέρει τα απαραίτητα αποτελέσματα. Έχει οδηγήσει σε κρίση τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με του παραγωγού αυτών των εξόχων απομακρυσμένων περιοχών με αυτή την αυστηρότατη δημοσιονομική επιθαρχία και του περιορισμού που του επιβάλλονται, ιδίω με το άνοιγμα των νέων αγορών και όλε τι συνέπειε τη κρίση που μόλι περιέγραψα. Ευχαριστούμε κύριε Φροντζούλικα για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να εκφράσω τη θετική μου άποψη, άρα και θα υπερψηφίσω ε, για αυτό το αποθεματικό για το 2015, διότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να στηρίξουμε περαιτέρω το γεωργικό τομέα. Και αυτό σε περίπτωση που προκύψει μια μείζον κρίση η οποία θα επηρεάσει τη γεωργική παραγωγή ή τη διανομή των γεωργικών προϊόντων με την ε, εφαρμογή αυτής της μείωσης των άμεσων ενισχύσεων στις αρχές ε, του κάθε έτους με τον μηχανισμό δημοσιονομικής πειθαρχίας. Ελπίζω να μην χρειαστεί βέβαια το αποθεματικό, αλλά αν τελικά χρειαστεί, πιστεύω ότι θα είναι ένα σημαντικό μέσο για τον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα. Και όλοι θα ωφεληθούμε. Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, πολύ σαφή όροι προποθέσει για του δικαιού. Θέλω να ευχαριστήσω τόσο τον εισηγητή και του Σκιώδη. Ευχαριστώ. πρόεδρε. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υποστήριξα ε, το ταμείο αυτό και βλέπω ότι υπάρχει η διαπροσέγγιση. Πολλά άλλα μέσα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διάθεσή τη σε ό,τι αφορά κάποιου γεωργού σε κάποια κράτη-μέλη. Γιατί τα πιο πολλά χρήματα δεν είναι πάντα η λύση. Χρειαζόμαστε πιο ελεύθερη, πιο αποδοτική ΚΑΠ που θα επιτρέψει να είναι ανταγωνιστική η γεωργία μα. Αυτή είναι η απάντηση. Το βασικό μου πρόβλημα όμως είναι η αδικία που υπάρχει στα μέσα χρηματοδότησης. Το όριο των 2.000 ευρώ σημαίνει ότι οι πιο μεγάλε χώρε θα πληρώσουν τα πιο πολλά. Τρία κρατημέλα θα πληρώσουν τίποτα. Πώς είναι αυτό το αλληλέγγυο. Αν είναι να υπάρξει ένα ταμείο ε, για την κρίση θα πρέπει να συνεισφέρουν όλοι οι γεωργοί και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει καν το ταμείο αυτό έτσι όπως έχει τα πράγματα όμως θα επιβαρυνθούν κάποιοι πιο πολύ από άλλους και έτσι τα βλέπουν σίγουρα τα πράγματα και οι γεωργοί στις, ε, στον Εμένο Βασίλειο ότι αυτοί θα πληρώσουν τους άλλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Κωστίν για δύο λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Επίτροπε. Εγώ τα αξιολογώ τα πράγματα λίγο διαφορετικά από το κύριο Ντάλτον. Πιστεύω ότι το εμπάργκο για τη Ρωσία σε καμία περίπτωση δεν προκλήθηκε από τους Γεωργούς και έχουμε σίγουρα καθήκον εδώ να βοηθήσουμε να συνδράμουμε και νομίζω ότι το εμπάρκο αυτό καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι το αποθεματικό κρίση στον τομέα της γεωργίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για παράδειγμα, ο κλάδος των απορκυπευτικών κατάφερε με τα ειδικά αυτά μέσα να απαλλαχθεί κάπως από την πίεση για την ε, Αυστρία. Αυτό σημαίνει εκατοντάδες ε, εκατομμύρια ευρώ για εξαγωγές σε τρίτες χώρες και έτσι ε, μείωση της πίεσης. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουν νόημα τα μέτρα αυτά σε εποχές κρίσης, αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω κατεπηγόντως το εξή ότι στο σημείο αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία, για παράδειγμα, για την ενημέρωση για τα μέτρα αυτά. Θα πρέπει να βελτιωθεί. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα το οποίο θα είναι αποτελεσματικό και γρήγορο θα πρέπει να υπάρχει όλο και πιο πολύ γραφειοκρατία σε τέτοιε περιπτώσει κρίση. Θα πρέπει να παρακαλέσω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σημείο αυτό να κάνει μια αξιολόγηση εκτεταμένη των μέτρων ενίσχυση. Να μην περιμένουμε την επόμενη κρίση για να βελτιώσουμε τα συστήματά μα σε Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίλυση των κρίσεων σε ό,τι αφορά και τον κατάλληλο προπολογισμό. Και κλείνοντα, θα ήθελα να πω πως η συνάδελφο Ριμπέρο το εξή για τον μικό κλάδο στι 31 Μαρτίου εξέπρεψε το σύστημα ε, επιδοτήσεων για, και ποσοστώσεων για το γάλα. Αυτό λοιπόν οδηγεί τους παραγωγούς σε μεγάλες προκλήσεις και του χρόνου θα αντιμετωπιστούν επιπλέον πιέσει στον τομέα γαλακτοκομικών. Κύριε Επιτροπέ, λοιπόν, σας παρακαλώ να κάνετε ό,τι μπορείτε προκειμένου να ενισχυθεί ο κλάδος των, της παραγωγής γαλακτοκομικών. Ευχαριστώ πολύ. Κάστρο για δύο λεπτά. Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Ο κανονισμός που θα ψηφίσουμε αύριο έχει να κάνει με μια ε, δημοσιονομική πειθαρχία, ο μαθηματικός υπολογισμός της Επιτροπής που θα δημιουργήσει ένα αποθεματικό αντιμετώπιση τη κρίση για το 2016 ορίζει ένα ποσοστό αναπροσαρμογή για τι άμεσε πληρωμέ του 2015. Η ομάδα μα θα υπερψηφίσει την πρόταση κανονισμού και την έκθεση του κ. Σικέρσκη, που ήδη την έχουμε εγκρίνει στην Επιτροπή Γεωργικών Υποθέσεων με την απλουστευμένη διαδικασία. Ωστόσο, η συζήτηση αυτή μα δίνει την ευκαιρία να υπογραμμίσουμε ότι ο μηχανισμό δημοσιονομική πειθαρχία είναι καρπό και αποτέλεσμα τη μείωση του προπολογισμού τη Γεωργία που από αποφασίστηκε στα πλαίσια τη μεταρρύθμιση 2014-2020 και δεν υπάρχει περιθώριο για να αντιμετωπίσουμε τι κρίσει που πλήττουν του γεωργού. Η κρίση όμω είναι κάτι που επαναλαμβάνεται διαρκώ ω φαινόμενο, όπω ήδη υπόθηκε. Το είδαμε με το ρωσικό εμπάργκο. Επιπλέον, οι τιμέ διαρκώς ε, είναι κειμενόμενες, όλο και περισσότερο μάλιστα μεταβάλλονται. Οι ίδιοι οι γεωργοί με τη μεταρρύθμιση του πρώτου πυλώνα της ΚΑΠ έχουν αναγκαστεί να πληρώσουν το τίμημα για αυτή την κρίση. Ε, με την προοπτική μιας μακράς περίοδου προσαρμογής θα πρέπει, Επίτροπε, να επινοήσουμε νέα μέτρα αντιμετώπιση της κρίσης, νέα και πιο ισχυρά, που να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα δίχτυ ασφαλείας για τους γεωργούς και να ε, τους επιτρέπουν να είναι ανταγωνιστικοί στη διεθνή αγορά χωρίς να φοβούνται. Επίτροπε, στην προηγούμενη προηγούμενη θητεία το Κοινοβούλιο είχε υποστηρίξει ότι η δημοσιονομική πειθαρχία θα πρέπει να επιβαρύνεται μόνο στους γεωργούς που λαμβάνουν πάνω από 5.000 ευρώ για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε περισσότερο τους μικροπαραγωγούς. Ωστόσο, δυστυχώς, το τελευταία συμφωνία το ε, όριο ρίστηκε στα 2.000 ευρώ. Εμείς συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι το όριο θα έπρεπε να είναι ανώτερο για να είμαστε δικαιότεροι και να μην μειωθούν οι πληρωμές προς τους μικρού παραγωγούς ε, αλλά να πληρώσουν αυτούς για τους οποίους μια μικρή μείωση της άμεσης πληρωμής τους από την ΚΑΠ δεν έχει σοβαρό αντίκτυπο στις δραστηριότητες τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαριάς. Την ώρα που ο Ντράγκη διαθέτει 1,1 τρισεκατομμύρια ευρώ για αγορά ιδιωτικού και δημοσίου χρέους, το ποσό των τετρακοσίων εκατομμυρίων ευρώ του αποθεματικού για την αντιμετώπιση κρίσεων στο γεωργικό τομέα είναι ψίχουλα για τους αγρότες της ελλάδας και της υπόλοιπης νότιας ευρώπης που πλήττονται από το ρωσικό εμπάργο και έχουν χάσει μέχρι σήμερα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. οι φτωχοποιημένοι από το μνημόνιο έλληνες αγρότες έχουν επίσης φέτος δοκιμαστεί και από τις καταστροφές στην παραγωγή τους λόγω των θεομηνιών που έπληξαν την πατρίδα μου ταυτόχρονα η φοροεπιδρομή που βιώνουν και φέτος οι έλληνες αγρότες με εντολή της τρόικας επεκτάθηκε παράνομα και στις κοινοτικές ενισχύσεις που λαμβάνουν. έτσι τα τελευταία πενταετία το εισόδημα των ελλήνων αγροτών μειώθηκε κατά 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ και οι φόροι που κατέβαλαν αυξήθηκαν κατά. 150%. για τους λόγους αυτούς πρέπει το ποσοστό αναπροσαρμογής δηλαδή το ποσοστό μείωσης που καθορίζει ο υποσυζήτηση κανονισμός να μην εφαρμοστεί στις ενισχύσεις που χορηγούνται στους έλληνες αγρότες αφού σε περίπτωση μη εξαίρεσης των ελλήνων αγροτών αυτό θα οδηγήσει σε νέα άδικη μείωση των εισοδημάτων τους. ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο καλός νομικός σχεδιασμός σίγουρα είναι δύσκολο έργο ε, σε οποιοδήποτε οργάνωση. Η κατάρτιση του προπολογισμού πρέπει σίγουρα να λαμβάνει υπόψη και την ανάγκη ε, ποιότητα ζωής για τους Ευρωπαίους πολίτες. Έχουμε λοιπόν την κατάρτιση του προπολογισμού του 2016 στο πλαίσιο του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Είναι πολύπλοκο εγχείρημα Έχουμε του όρου της κοινή γεωργική πολιτικής, έχουμε τον κανονισμό για αυτό το αποθεματικό για την αντιμετώπιση κρίσεων. Το ποσό του αποθεματικού που θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο σχέδιο περιπολογισμού για το 2016 είναι 441,6 εκατομμύρια ευρώ και θα αντισταθμιστεί από τις άμεσες ενισχύσεις που καταβάλλονται σε γεωργούς ε, που παίρνουν πάνω από 2.000. Έχουμε λοιπόν μείωση ε, της τάξης του 1,393% δεν θα εφαρμοστεί αυτή η μείωση για Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία. Η Ευρωπαϊκή Γεωργία ε, έχει αντιμετωπίσει απώλειες λόγω πολιτικών αποφάσεων όπως ε, το ρωσικό εμπάργκο. Πρόκειται για μια κρίση που δεν την προκάλεσαν οι ίδιοι οι αγρότες. Πιστεύω λοιπόν ότι οι αποζημιώσεις στους αγρότες δεν θα πρέπει να καταβάλλονται από το γεωργικό προϋπολογισμό, αλλά από άλλες πηγές. Το αποθεματικό για το οποίο συζητούμε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ε, προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για κρίσεις που θα προκαλούνται στο γεωργικό τομέα. Καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν να εξασφαλίσει και αποζημίωση ε, των παραγωγών γάλακτος διακόπτεται. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως και οι συνάδελφοι από την ομάδα και εγώ συμφωνώ με όσα υπόθηκαν για την κρίση σε ό,τι αφορά το αποθεματικό και όσα προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ομολογώ ότι είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες οι προτάσεις. Θα ήθελα όμως να επιστήσω την προσοχή σας στο εξή. Τι γίνεται στην Ουγγαρία. Είναι αντιφατικά τα μηνύματα που αποστέλλονται στις άμεσες επιδοτήσεις ε, βλέπουμε και στα διάφορα ταμεία αποσμίωσης ότι οι ολιγάρχες και οι πολιτικοί φίλοι που παίρνουν ε, τα χρήματα τελικά. Αυτό φυσικά είναι δύσκολο να αποδειχτεί, αλλά είναι χαρακτηριστικό των διεφθαρμένων ε, κυβερνήσεων. Τις τελευταίες ημέρες συνελήφθησαν δύο άτομα και 100% διαπιστώνουμε ότι στην Ουγγαρία τα... οι ενισχύσεις πάνε στους ολιγάρχες και η Ουγγρική κυβέρνηση υποστηρίζει αυτούς τους ολιγάρχες. Καλωσορίζω σε κάθε περίπτωση την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τότε να μπορεί να ελέγχονται ποιος λαμβάνει την υποστηρίξη. Θα πω ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο τομέας αυτός ε, σε περίπτωση κρίσης πρέπει να προστατεύεται. Είναι σημαντικό να υπάρχει αποθεματικό όταν μιλάμε για επιστημιστική ασφάλεια. Πρέπει λοιπόν για τις έκτατε ανάγκες, όπως σήμερα, που έχουν γίνει και ο κανόνα και όχι εξαιρέσει για το ειδικό τομέα, να προβλεφθεί. Ο τομέας δοκιμάζεται από το ρωσικό εμπάργο και τις ε, ποσοστώσεις του γάλακτο βλέπουμε τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και τη διεθνή κρίση που υπάρχει. Το απαθηματικό λοιπόν που προβλέπεται για το σχέδιο προπολογισμού του 2016 από την Επιτροπή σε 441,6 εκατομμύρια ευρώ ε, με τρέχουσες τιμές είναι σημαντικό. Θα πρέπει όμως να χρησιμοποιείται μόνο εφόσον χρειάζεται και δεν είναι αυτό μια ε, αποτελεσματική οριστική λύση για τον γεωργικό τομέα. Ο κόσμος της γεωργίας ε, έχει πληρώσει το τίμημα για τις διάφορες κρίσεις. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επίτροπο Χόγκαν, το οποίο εκτιμώ τις πρωτοβουλίες, θα πρέπει να βρει δικαιότερε λύσεις με το πρόθεσμα. Ευχαριστούμε ο κύριος Άγνιου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το θέμα στο οποίο συμφωνούμε όλοι είναι ότι δεν υπάρχει σαφήνεια για τους κανόνες από τον Επίτροπο. Βλέπω τον κύριο Χόγκαν ε, στρέφεται να με κοιτάξει και αυτό με το λακεύει. Αλλά ήδη 15% ε, μείωση στις πληρωμές τους έχουν ε, οι Ιρλανδοί Γεωργοί λόγω της αδυναμίας του ευρώ. Γιατί είναι τόσο αδύναμο. Διότι ουσιαστικά το χρησιμοποιούν χώρες που δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να συμμετέχουν στο κοινό νόμισμα. Αυτό ε, ίσως να μην είναι μια θεόσταλτη απόφαση, αλλά είναι κάτι που το αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα θεσμικό όργανο που λειτουργεί ως θεότητα και θα μπορούσε κανείς να την ε, περιγράψει και έτσι. Το αποθεματικό αυτό λοιπόν υποκαθιστά αυτό που ονομαζόταν ε, το πράσινο περιθώριο, αυτό που μπορούσε να ε, ενεργοποιήσει πληρωμές στους γεωργούς που είχαν χάσει ευκαιρίες εξαγωγών και στην περίπτωση που είχαν μειωθεί οι, εθνικές, οι τιμές σε εθνικό επίπεδο λόγω της αδυναμίας του ευρώ. Αυτό είναι ένα επιχείρημα για το Ηνωμένο Βασίλειο να μην συμμετάσχει στο ευρώ ούτως ή άλλως. Και ξέρετε ότι αν το είχαμε κάνει κύριε Επίτροπε, οι φορολογούμενοι θα είχαν στραγγαλιστεί και θα έπρεπε να πληρώνουν και να χρηματοδοτούν την ΚΑΠ. Είναι λοιπόν πολύ βολικό να ξέχουν τα κρατημέλη ότι ο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα από του βασικού συνεισφέροντε στην ε, ΚΑΠ. Άλλοι φορολογούμενοι θέλουν να ξέρουν ότι τα χρήματά του τουλάχιστον χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν την εγχώρια παραγωγή και τα εγχώρια γεωργικά προϊόντα και όχι κάτι πολύ απόμακρο. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Επίτροπε θα ήθελα να τοποθετηθείτε συγκεκριμένα επί του θέματος αυτού. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ απόψει Ευχαριστούμε. Και τώρα στη διαδικασία ΚΑΤΣ Eye προσέλκυση τη προσοχή του Προέδρου. Έχουμε τέσσερι συναδέλφου που έχουν ζητήσει τον λόγο και θα δώσω τον λόγο σε όλου. Πρώτα απ' όλα, ο κ. Γκλέζο. Αγαπητοί συνάδελφοι, α μην στρουθοκαμιλίζουμε και α μην ρίχνουμε την αιτία της κατάστασης των, αγροτών, των μας στο ρωσικό εμπάργκο. Πριν από το ρωσικό εμπάργκο υπήρξε το εμπάργκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος το χειρών αδίκων. Πρώτος ήρξατο η χειρων αδικων πρωτος ήρξα το ευρωπαικη ενωση Και αναμφισβήτητα το προνοεί είναι χρήσιμο. Πρέπει να υπάρχει ένα ταμείο για την αντιμετώπιση των ε, θεομηνιών. Αλλά ειδικά για την ελλάδα θέλω να σημειώσω το γεγονός ότι πέρα από την οικονομική κρίση που δεν την προκάλεσαν οι έλληνες αγρότες ε, ούτε η πολιτική των θεσμών απέναντι στην αγροτική μας οικονομία είναι τρομερή. Δεν θέλουν να αναπτυχθεί η αγροτική οικονομία στην Ελλάδα. Δεν μας θέλουν ούτε βιομηχανική χώρα, δεν μας θέλουν ούτε ε, ε, αξιοποίηση των ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μας θέλουν ένα θέρετρο. Ένα μεγάλο ξενοδοχείο θέλουν την Ελλάδα. Domnul ε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Στηρίζω αυτό το ποσοστό αναπροσαρμογής ε, για τις άμεσες ενισχύσεις το 2015 που θα εφαρμοστεί το 2016 και στην προκειμένη περίπτωση είναι γεγονός ότι αν θέλουμε να δώσουμε κάτι πρέπει να το πάρουμε από κάπου αλλού. Γι' αυτό και χρειάζεται η σωστή εποπτεία για την ε, διάθεση αυτών των κονδυλίων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για μετριασμό των επιπτώσεων ε, μια ενδεχόμενη κρίση. Γι' αυτό τα κριτήρια που θα εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, κατανομή αυτών των κονδύλων θα πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρα, σταθμισμένα και να συνοδεύονται από αποτελεσματική εποπτεία, όπως είπα. Δεν θα πρέπει να προκύψει μια κατάσταση όπου θα πρέπει να συζητούμε τις ατασταλίες και παρατυπίες του παρελθόντος. Γι' αυτό η αποτελεσματική χρήση και η τακτική χρήση των ε, κονδυλίων είναι απαραίτητη. Thank ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι γεγονός ότι η κρίση και η κρίση χτυπών τον κόσμο. Χρειάζονται λοιπόν αποθεματικά. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε χρήματα σε τέτοιο χαμηλό επίπεδο. Υπάρχουν ε, κατεπίγουσες ε, περιπτώσεις ανάγκης και θα πρέπει σε τοπικό επίπεδο τα κράτη-μέλη να έχουν δυνατότητε. Τα κράτη-μέλη έχουν τις λύσεις. Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε. Και για 500 εκατομμύρια άτομα από το βορρά μέχρι τη Σαρδενία να έχουμε τις ίδιες λύσεις. Πότε θα καταλάβατε ότι το μεγάλο ή μεγάλη κλίμακα είναι κάτι αρνητικό. Το μικρό είναι όμορφο και το, σε το τοπικό επίπεδο τα πράγματα γίνονται πραγματικά όπως πρέπει τα πράγματα. Αυτό επιθυμούμε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Μορβάη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άξιο ότι με κύριε Επίτροπε. Στα συγκεκριμένα ζητήματα θα ήθελα να σας παρακαλέσω για κατεπίγουσα βοήθεια. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται στην Ουγγαρία. Υπάρχει ένα εθνικό πάρκο το οποίο επισκέφθηκα αυτό το Σαββατοκυριακό και έμαθα πραγματικά συγκλονιστικά πράγματα τα οποία θα ήθελα να σας κοινοποιήσω. 15 χιλιόμετρα σε έκταση 15 χιλιόμετρων σε μεγάλες σε παιδιάδες δεν υπάρχει ούτε ένα ούτε ένα ζώο. Γιατί, γιατί τα ζώα τα κρατάνε στους ε, σταύλους. και οι γέργοι έχουν χάσει μεγάλο μέρος των εισοδημάτων τους και λόγω της διαφθοράς πτωχεύουν και αν πάτε εκεί θα δείτε ότι οι άνθρωποι που ζουν εκεί, που ζούσαν εκεί δεν ξέρουν τίποτα, δεν, δεν έχουν καμία γνώση στα γεωργικά ζητήματα. Θέλουν μόνο τι επιδοτήσει να πάρουν. Θα πρέπει να ελέγξετε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο τώρα στον Επίτροπο Χόγκαν. Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλα τους βουλευτές που συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή. Να ευχαριστήσω και ιδιαίτερα τον κύριο Σικέρσκη τον εισηγητή που εργάστηκε για την ε, έκθεση αυτή. Θα ήθελα να μιλήσω για την τελευταία μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΠ και να επικρατήσω την ύπαρξη ενός ταμείου αποθεματικού. Αυτό καταδεικνύει την αλληλεγγύη με την κοινότητα των γεωργών και καλλιεργητών σε περιπτώσεις και περιόδους κρίσης. Καλωσορίζω λοιπόν τα μέτρα που λήφθησαν το 2015. Το αποθεματικό για την κρίση είναι η αλληλεγγύη σε δράση. Αυτό του ταμείου, όπως σας είπα, κρηματοδοτείται από τις υφιστάμενους πόρους της ε, κοινότητα των Γεωργών. Πολλοί αναφέρθηκαν στο ρωσικό εμπάργκο. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Οκτώβριο έκανε μία πρόταση που θα είχε χρησιμοποιήσει αυτό το ταμείο 413 εκατομμυρίων ευρώ. Και τον Νοέμβριο ε, άλλαξε η απόφαση αυτή προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από άλλες πηγές το ταμείο αυτό. και στην περίπτωση αυτή θα είχε κοστίσει 350 εκατομμύρια το Ταμείο, χωρίς να αναφερθεί το Ταμείο Κρίσης. Ο κύριος Δαντών μίλησε για το Ταμείο αυτό, αλλά έχετε ξεχάσει τις αποφάσεις που ελήφθησαν το Νοέμβριο για να αλλάξουν οι αποφάσεις και να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Τζεωτζίεβα που έδειξε μεγάλη κατανόηση σε ό,τι αφορά το χειρίο Κρέα. να πω το γεγονός ότι αναγνωρίζουμε τις δυσκολίε για πολλές χώρες. Το αποθεματικό άνοιξε για 10 εβδομάδε και σίγουρα σταθεροποιεί την κατάσταση για πολλούς παραγωγού χειρίου κρέατο. Επίση ε, ανοίγει κάποιε αγορέ πρόσθετες εξαγωγών για να αντισταθμιστούν ε, οι συνέπειε του εμπάρκου, όπως για παράδειγμα οι Φιλεπίνε, 73% τώρα των ε, προϊόντων που πήγαιναν στην Ρωσία απορροφούνται σε άλλε αγορέ. Άρα, στον τομέα του χειριοκρέατος βλέπουμε πώς λειτουργεί η αλληλεγγύη σε ό,τι αφορά την επιθεαρχία και την προσαρμογή. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι εξαιρούνται οι μικροί ε, γεωργοί από το όριο των 2.000 ευρώ και σε ό,τι αφορά αυτά που είπε ο κ. Άσχουερθ ότι πολλοί γεωργοί στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της δομής του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα πρέπει να πληρώσουν αυτή την εισφορά. Αυτό όντω αποτυπώνει την, την πραγματικότητα ότι οι μικρομεσαίοι παραγωγοί έχουν την ικανότητα και την δυνατότητα να πληρώσουν τα, τις φορές αυτές. Ο κύριος Άγνιο έκανε κάποια άλλα σχόλια για το Ενωμένο Βασίλειο αλλά θα ξέρει καλά ότι όταν ψάχνει κανείς 25 δισεκατομμύρια που αυτό είναι το ποσό που πληρώνουμε στους ε, αγρότες ε, του Ηνωμένου Βασιλείου, τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι λοιπόν γενναιόδορη η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τους ε, αγρότες του Ηνωμένου Βασιλείου και η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα θα είναι πιο γενναιόδοροι προς του Αγρότε του Ηνωμένου Βασιλείου από ότι θα είναι η ίδια η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Καλωσορίζω λοιπόν την πρόταση αυτή και προσβλέπω σε μια θετική ψηφοφορία αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή Σικέρσκη. E, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επιτροπέ, κυρίε και κύριοι. Πρόκειται για μια τεχνική έκθεση και η συζήτηση ήταν άκρο τεχνική, με ευγνώμους όλους του συναδέλφους. Η ταχεία διαδικασία για την έγκριση του εν λόγω εγγράφου σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη βαθμό συμφωνίας ε, μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Κομισιών. Το οποίο είναι σημαντικό όταν χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε επίγουσες καταστάσεις. Ε, έγινε λόγος για αλληλεγγύη και ναι πράγματι σχεδόν όλοι ε, πλην των πολύ μικρών συνεισφέρουν σε αυτό το αποθεματικό, σε αυτό το ταμείο το οποίο θα το χρησιμοποιούν ε, όσοι πλήττονται από την κρίση. Άρα πράγματι η αλληλεγγύη παίζει σημαντικό ρόλο. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η γεωργία είναι ένας ε, ιδιαίτερος τομέας. Ξαρτάται από τον καιρό, από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά και από την διεθνή κατάσταση. Επομένως, χρειαζόμαστε μέσα που ίσως να μην δημιουργούνται πάντοτε από την ελεύθερη αγορά, η οποία χρειάζεται ένα είδος υποστήριξης για την αντιμετώπιση ορισμένων κρίσεων. Μία μείζωνα δυναμία της μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής είναι ο περιορισμός ε, της παρέμβασης στην αγορά. Το είπα και προηγουμένως. Οι παρεμβάσεις περιορίστηκαν, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σίγουρα χρειάζεται μια καλή διαχείριση. Όμως, εν γέννη, έχουμε λιγότερα κονδύλια για τη γεωργική πολιτική και για τη γεωργία. Δεν θα πρέπει όμως να υποστηρίζουμε ότι την κρίση την προκάλεσε η γεωργική πολιτική γιατί δεν λαμβάνουν στήριξη και ενίσχυση μόνο οι γεωργοί, αλλά και οι καταναλωτές ωφελούνται από ε, τις, τα μέτρα αυτά, καθότι είναι πιο φθηνά τα τρόφιμα. Αυτά και ευχαριστώ και τον Επίτροπο για τη συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση και αύριο θα γίνει η ψηφοφορία. Μάλιστα. Επόμενο σημείο στην εμπειρία διατάξη έχουμε την έκθεση της κυρίας